Il Presidente. Acceso. Buongiorno colleghe e colleghi. Καλημέρα συνάδελφοι. Στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε την ε, ε, έκθεση Κιν Κακάλ ε, σχετικά με την ε, ουσιαστική εφαρμογή των θεμελιών δικαιωμάτων μετά την αριστερή ισχύ ε, της Συνθήκης Λισαβόνας. Το λόγο έχει η συγγήτρια για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε,